Welcome ήρθατε συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Ετοιμαστείτε για τουλάχιστον μια μισή ώρα ψηφοφορία. Uh, Λυπάμαι πολύ. Όμω δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Πρέπει να γίνουν αυτέ τι ψηφοφορίε. Ξεκινούμε με μία δοκιμή. Μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Παρακαλώ να βάλετε τις κάρτες σας. Δεν ξέρω, είστε δυσαρεστημένοι από τις θερινές διακοπές. Γιατί ξέρω ότι πόσο πολύ αγαπάτε την Ήτρια και δεν θέλετε να φύγετε λόγω διακοπών.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 στην πρώτη πρόταση για την ψήξη και θέρμανση. Ο Άνταμ Γέρεκ είναι εισηγητής. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. την 102. I open the vote. I close the vote. Accepted. Accepted. Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 117. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 118. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά. απόχέ απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά. αποχέ απορρίπτεται. 125 υπέρ. Κατά. απόχέ απορρίπτεται. 127 υπέρ. Κατά. αποχέ. εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. απόχέ απορρίπτεται. 129 υπέρ κατά, Αποχέ απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, Αποχέ αποχές Ένδυ NV5 υπέρ, κατά, αποχέ εγκρίνεται. 144 υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. 140 υπέρ, κατά, Αποχέ απορρίπτεται. 158 εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 166 υπέρ. Απορρίπτεται. 168 δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 168 δεύτερο τμήμα. Πέρας. 173 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 179 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 183 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 198 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 201 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. NV25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. NV15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. NV2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 224 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 2.25 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.27 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.29 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.47 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.48 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2.49 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.52 δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 2.61 υπέρ, κατά αποχές Εγκρίνεται. 262 υπέρ. 262 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 258 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 263 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 264 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται αυτή τη φορά. 265, 266 είναι ταυτόσιμες. ψηφίες μου από κοινού. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 267 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 269 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 268 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 285 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 286 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 290 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. NB34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 291 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 293 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 294 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Τη 294 ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 292 υπέρ. Κατά. Ας ελέγξουμε. 2.92. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 2.96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 300 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 301 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 302 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 303 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 304 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 305 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 306 υπέρ, Κατά. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 406. I close the Εγκρίνεται. Ο πρόεδρο λέει ότι υπάρχει δυσκολία με τη διερμηνία. Μήπω να μ' ακούτε στα αγγλικά, λέει ο πρόεδρο. Οι διερμηνεί απλώ δεν έχουν το κείμενο των ψηφοφοριών. Αυτό είναι το πρόβλημα. I've got a, written, written form. Please be slower. Μου έχουν στείλει σημείωμα οι διερμηνεί, λέει ο πρόεδρο, αν μπορείτε να διαβάζετε πιο αργά. So, 306 was accepted. 306 was accepted. I, I will be a bit slower. Θα είμαι λίγο πιο αργός. 307 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 308 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 318 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 319 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 320 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. ΕΝΒΙ 30 υπέρ. Κατά αποχές. Ας ελέγξουμε. Την ΕΝΒΙ 30 I close the vote. Accepted. Accepted. Compromise 16 in favor. Εγκρίνεται. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 329 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 330 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπτεται. 331 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 335 υπέρ. Κατά. Κατά. 335 και πάλι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 336 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 337 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 338 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 339 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε τώρα. 339. 339. I open the vote. I... Ένας ψηφοφορίας. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Uh, 341 in favor. 341 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.42 υπέρ, κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Την 3.42. Accepted. Εγκρίνεται. 3.44 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εγκρίνεται 3.44. 3.45 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρεις τροπολογίες μαζί. 7, 8, 9. Υπέρ. κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίες. εγκρίνεται. 3.50. Όχι, συγγνώμη, συμβαστική 21. Ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3-5-7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3-5-5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3-59 υπέρ κατά απορρίπτεται υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 361 υπέρ Κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. 361. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 363. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 362. Υπέρ. Κατά. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πέρα Εγκρίνεται. 364. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 366. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 368. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 369. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 370 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ένβη 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. συμβιβαστική 23α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 370 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 373 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 376 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 377 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 379 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 383 υπέρ κατά Αναποφάσου σας βλέπω. Ξανά. Τροπολογία 383 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 384 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 387 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 25α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 396 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 398 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 400 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 402 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 406 υπέρ κατά να ελέγξουμε για την 406 ψηφίζουμε τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται 407 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 408 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 420 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 423 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 424 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 426 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 427 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 26B υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 428 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4.30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4.31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4.34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 435 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 442 υπέρ κατά αποχές ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 442. Ψηφίστε παρακαλώ. I close the vote. Accepted. Εγκρίνεται. 4.43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 4.43 παρακαλώ. Ψηφίστε. I close the vote. Oh, see. Rejected. Απορρίπτεται. 4-4-4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4-45 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4-46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. NV22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. NV39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία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 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική β α νέο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές 49, ε, απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Ι e. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Κάτι, κάτι δεν πάει πολύ καλά με την ε, ψηφοφορία εδώ. Δεν κατάλαβα ακριβώ. Λοιπόν, τροπολογία 59. Ψηφίστε. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά είναι λίγο περίπλοκο. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. I close the vote. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 61 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 66 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 84 παρακαλώ. Τροπολογία 84 πέρα τη ψηφοφορία εγκρίνεται. Τροπολογία 85 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση επί της ε, τροπολογίας 93 93 Πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία διονομαστικής κλίσεως Άρχεται η ψηφοφορία για, επί του συνόλου της προτάσεως όσο έχει τροποποιηθεί. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. 47 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος εναντίον, 8 αποχές. Πολύ καλό αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι ο προϋπολογισμός. Κύριε Κάρενς, πριν ψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα ε, για τον προϋπολογισμό 2017 όλα τα τμήματα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι διαδικαστικό. Στις τροπολογίες 35 και 36 ε, υπάρχει αίτημα του κυρίου Μαρινέσκου ότι μπορούν να ψηφιστούν από κοινού. Πρόκειται για πιλωτικά προγράμματα ε, ε, για το διάστημα και η πρόταση είναι οι 35 και οι 36 να ψηφιστούν από κοινού. Πολύ ωραία. Θα το συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα θα πρέπει να δείξετε ιδιαίτερη ε, υπομονή γιατί έχουμε 45 σελίδες ψηφοφορίας. Έχετε όλοι τον κατάλογο ψηφοφορίας, ψηφοφορίας. Ε? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε όλοι τον ίδιο μορφότυπο, 45 σελίδες, για να μπορούμε να ακολουθούμε όλοι ε, το ίδιο κείμενο. Εάν δεν έχετε τον ίδιο μορφότυπο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα, αλλά θα πρέπει να το ξέρω, γιατί, ε, α, οκ, okay, το κατάλαβα, άλλοι έχουμε 40 σελίδες, άλλοι 45, άλλοι παραπάνω, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ας ξεκινήσουμε.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 κατά αποχές εγκρίνονται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 όχι 41 41 υπέρ 41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 69 μία ακόμα φορά υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Η ε, ηλεκτρονική επαλήθευση από τις τροπολογίες 72. Ηλεκτρονική, ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν. Πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, όχι, καλύτερα να ελέγξουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν από τις τροπολογίες 73 και πέρας της ψηφοφορίας αποδεκτή. Τροπολογία 75 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 77 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά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 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 96 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 98 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 99 υπέρ. Κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 106 ε, ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 106 ε, πέρας της ψηφοφορίας και απερίφθη 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά νομίζω και εδώ η ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 109 άρχεται πέρας της ψηφοφορίας και απερίφθη 110 Α, απερίφθη 110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 Ελέγχουμε το αποτέλεσμα για την 130 πέρα στις πληροφορίες. Απερίφθη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ που μου το υποδείξατε. 131 υπέρ κατά αποχές. Απερίφθη 132 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ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 could be would be much... Συνάδελφοι, θα ήταν σίγουρα πολύ πιο βολικό για μένα, αλλά σε σχέση και με την ε, παρελθοντική μας εμπειρία και για λόγους διαφάνειας για την πόλη εκθέσεων, ξέρουμε κιόλας ότι κάποιοι συνάδελφοι πολύ συχνά καταψηφίζουν έχουμε ευρύτατη πλειοψηφία υπέρ της αποδοχής. Ορισμένοι συνάδελφοι όμως καταψηφίζουν. Γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να πούμε ότι υπάρχει κάτι σαν συμβαστική τροπολογία στις επιμέρους γραμμές υπολογισμού. Ας λάβουμε λοιπόν υπόψη την εμπειρία μας από προηγούμενες ψηφοφορίες στην Ήτρε. Πάντα τις ψηφίζουμε όλες. So I'm sorry. 152. 152. 152 152. υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 153 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 155 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ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 Ελέγχουμε την 194. Πέρας. Απορρίπτεται. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. Με προφανή τρόπο. Εσείς ως συντονιστές δεν μπορείτε να κάνετε κι αλλιώς. Πρέπει να το σηκώσετε το χέρι. Αλλά και οι υπόλοιποι συναδέλφοι παρακαλώ. Σηκώνετε τα χέρια σας γιατί δεν τα βλέπω. 195 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 6 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται είστε εντελώ μόνος τώρα 7 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά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 Τη 237. We check voting. The voting. I close voting. Is rejected. Απορρίπτεται. 2.38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελπίζω να εγκρίνονται. Οι σοσιαλιστές δεν ψήφισαν καθόλου. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 45 περ. κατά αποχές εγκρίνεται 46 περ. κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 250 υπέρ κατά ας ελέγξουμε 250. We check 250. 250 ελέγχουμε. I close the vote. Is rejected. 200... Απορρίπτεται. 251. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53. Υπέρ. Κατά αποχές. 2.53, ελέγχουμε. Has anybody voted? I close the vote. Is rejected. 254. Απορρίπτεται. 254 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελπίζω να εγκρίνεται. Το ΕΛΚ δεν ψήφισε. 2.55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.57 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.58 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.59 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 2.60 υπέρ.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 ηλεκτρονικά. Πέρας. 43 υπέρ 8 κατά 7 αποχές. Επιβεβαιώνουμε εκ νέου τη γνωμοδότηση για τις γραμμές προπολογισμού τελική ψηφοφορία και πάλι με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας. 43 υπέρ 8 κατά 5 αποχές. Thank you very much, colleagues. Ευχαριστώ συναδελφοί για την υπομονή σας. Πάμε σε άλλες δύο ψηφοφορίες τώρα. Ευτυχώς όμως θα είναι πολύ σύντομες. Μία ώρα. Εξαιρετικά. Συγχαρητήρια. Σχέδιο έκθεση για τι ευρωπαϊκέ στατιστικέ όσον αφορά τι τιμέ φυσικού αερίου και ηλεκτρική ενέργεια. Η, η συγκίτριά μα, κυρία Κάπελ, έχει καταλήξει σε ένα σχέδιο κειμένου με το Συμβούλιο. Τα συμφωνία. Τελικό κείμενο. Ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τώρα. Πέρας της ψηφοφορίας. 31 υπέρ, 8 κατά, 3 εποχές. Συγχαρητήρια. Πάμε σε μια ακόμη ψηφοφορία. Συμβολή της Επιτροπής Ήτρε στο ψήφισμα Τσέμβη για την COP22, τη συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον, που θα γίνει στο Μαρόκο, στο Μαρακές, στην Αφρική αυτή τη φορά. Σοφορία για το συμβαστικό κείμενο. Ηλεκτρονική σοφορία η οποία ξεκινά τώρα. Πέρασε φοφορίες. 51 υπέρ, 3 κατά, Τέσσερις αποχές. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους. Και ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες. Στην ώρα μας. Από ό,τι βλέπω, μην πω και λίγο νωρίτερα. Ωραία. Καθώς θα φεύγετε λοιπόν, όσοι φεύγετε από την αίθουσα, σας εύχομαι καλές διακοπές αν και θα προτιμούσα και θα σας παρακαλούσα να μείνετε για άλλη μια μισή ώρα. Τίποτα άλλο δεν θα σας πω, μόνο να σας παρακαλέσω για την επόμενη μια μισή ώρα για να συζητήσουμε με τον Επίτροπο μας. Τον Επίτροπο για ζητήματα έρευνας, επιστήμης και κοινοτομίας. ο κύριος Κάρλος Μοέντας έρχεται. Βλέπω ότι βιάζεστε να φύγετε για διακοπές. Τι να κάνω εγώ. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Επίτροπε, σας καλωσορίζουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Χαιρόμαστε πολύ που σας φιλοξενούμε άλλη μια φορά. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές να συζητήσουμε μαζί σας κάποια σημαντικά θέματα στα, στον τομέα της ε, έρευνας, επιστήμης και της κοινοτομίας και να συζητήσουμε και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις που έχετε καταθέσει. Πρώτα απ' όλα, στο, το, στο Συμβούλιο το ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας ε, και τα πορίσματα αυτού, νέα βήματα, επόμενα βήματα στο ορίζοντα 2020 η έκθεση της κυρίας Σολέδα Καμπεθών από τους σοσιαλιστές θα ψηφιστεί τον Ιούλιο του 2017 και επίσης σκοπεύουμε να κάνουμε και δύο αποστολές διερευνητικές στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Όσον αφορά το Ευρωπαϊκό cloud έχουμε και εισηγητή για αυτό το θέμα, για την δημιουργία μιας ανταγωνιστικής οικονομίας δεδομένων και γνώσης στην Ευρώπη. Παρ' αυτά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πραγματικά γιατί να σας συγχαρώ κι εγώ για... ή δεν ξέρω, να σας συγχαρώ ή όχι. Όχι, πάση περιπτώσει σας συγχαίρω για το αποτέλεσμα που έφερε η Εθνική Πορτογαλία ε, την Κυριακή στο Παρίσι. Όλοι, να συγχαρώ όλους τους συναδέλφους από την Πορτοκαλία. Έναν επίτροπο έχετε, αλλά έχετε και τον μοναδικό πρωταθλητή Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μοέδα στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου. Που είναι σημαντικό θέμα και για τις δύο πλευρές, και για το Κοινοβούλιο και για την ε, Κομισιόν. Έχουμε βεβαίως κοινού στόχους, αλλά οι συζητήσεις γίνονται μεταξύ δύο μερών. Κύριε ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα καλά σας λόγια. Ήταν πραγματικά μια πολύ συγκινητική στιγμή η βραδιά της Κυριακής και ήμουν και εγώ πολύ περήφανος για τη χώρα μου. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ στο πλαίσιο αυτού του διαρθρωμένου διαλόγου για να σας ενημερώσω για τα τρία ε, κύρια θέματα που θα καλύψω τα επόμενα ε, ε, λεπτά. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομία, το Open Cloud και το Horizon 2020. Ξεκινήσουμε με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομία. Να πω πρώτα απ' όλα ότι ευχαριστώ όλους σας για τις επικοδομητικές συζητήσεις που έχω κάνει με, μονομένα μέλη της Επιτροπής Ήτρε για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε στον τομέα της κοινοτομίας. Και πραγματικά μεγάλη δύναμη και ενθουσιασμό μου παρέχουν οι δικές σας ιδέες και γνώμες. Ο Ορίζοντας 2020 είναι το πρώτο πρόγραμμα πλαίσιο που αφορά την καινοτομία και την έρευνα και εισήγαγε νέες ε, ε, νέα εργαλεία, τα χρηματοπιστωτικά, τα δημοσιονομικά εργαλεία. Και η υψηλή συμμετοχή διαφόρων φορέων δείχνει ότι τα πάμε καλά. Όμως πρέπει να πω ότι στον τομέα της κοινοτομίας χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ορατότητα, χρειάζεται να αποδείξουμε τις θετικές επιπτώσεις που έχει η κοινοτομία στους διάφορους τομείς και αυτό που βλέπουμε είναι ότι πολλές από τις ε, καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νεοπαγείς εταιρείε, ακόμη δεν έλκονται πολύ από τα δικά μας προγράμματα. Βλέπω δηλαδή ότι κάποιες ε, από αυτές τις εταιρείε δεν γνωρίζουν καν τα προγράμματα μας και παρά την ε, επιστημονική δύναμη και ισχύ που έχει η Ευρώπη είμαστε ακόμα πίσω σε σχέση με τις ΙΠΑ και την ε, Ιαπωνία προκειμένου να καλύπτουν οι δικές μας εταιρείες σε αυτό το τομέα της καινοτομίας. Και η αλήθεια είναι ότι πολλές από τις νέες ε, καινοτόμες δικές μας επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν καν για το τι υποστήριξη μπορούν να λάβουν από ευρωπαϊκής πλευράς. Και όταν, το όταν γνωρίζουν τα προγράμματα αυτά, τα θεωρούν πολύ γραφειοκρατικά ή πολύ περίπλοκα. Οπότε πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους φορείς καινοτομίες νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε κάποιες αλλαγές και γι' αυτό τον χρόνο πέρσι προτείναμε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας. Πρώτα απ' όλα όμως να ξεκαθαρίσω προς κάθε πλευρά και να το κάνω και εδώ ότι χρειάζεται να καθορίσουμε τις παραμέτρους αυτής της συζήτησης. Και όπως έχω ξαναπώ, ε, σκοπός μας δεν είναι να δημιουργήσουμε νέα θεσμικά όργανα, το επαναλαμβάνω λοιπόν. Δεν θέλουμε λοιπόν να προσθέσουμε επιπλέον στρώματα περιπλοκότητας ή γραφειοκρατίας. Το αντίθετο θέλουμε να Άρα, σκοπός μας δεν είναι απλά να αλλάξουμε προϋπολογισμούς από την έρευνα στην κοινοτομία. Όχι. Σκοπός μας είναι πώς θα μπορούσαμε να απλουστεύσουμε και να ε, ενισχύσουμε την υποστήριξή μας προς την ε, καινοτομία. Δεύτερον, στο πλαίσιο αυτού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, εγώ είμαι πρόθυμος και έτοιμος να συνεργαστώ με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Θα συνεργαστούμε λοιπόν με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Έρευνας. Έχουμε ήδη ε, κάνει συζητήσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου και μου έχουν εκφράσει και τα μέλη αυτού ότι ενδιαφέρει, τα ενδιαφέρει και εκείνο η ενίσχυση της κοινοτομίας. Επίσης πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα κονδύλια τα δικά μας θα δρουν συμπληρωματικά προς τα εθνικά κονδύλια. Πώς θα μπορούσαμε δηλαδή να προσελκύσουμε ιδιωτικά κεφάλαια και πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε λοιπόν καταθέσει κάποιες βασικές ιδέες και νομίζω ότι είχαμε ε, πολύ καλές απαντήσεις μέχρι στιγμής. Άνω των χιλίων απαντήσεων έχουμε λάβει, αλλά έχουμε δει και 100 ε, εργασίες, μελέτες για αυτό το θέμα. Έγγραφα, θέσεις δηλαδή, από διάφορους ανθρώπους και διάφορους, διάφορες πλευρές. Όταν ξεκινήσαμε ε, δεν περιμέναμε να ξεπεράσουμε ούτε καν τις 100 απαντήσεις. Τελικά όμως λάβαμε χίλιες. Αυτά τα έγγραφα είναι πολύ σημαντικά για μας προκειμένου να ε, σχηματίσουμε μια εικόνα για το ποιε είναι οι επιθυμίες των ανθρώπων. Και νομίζω ότι τα μηνύματα είναι σαφή. Το πρώτο είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι πιο ανοιχτή προς την καινοτομία. Να αναλαμβάνει περισσότερους κινδύνους, περισσότερο ρίσκο και να είναι πιο ανοιχτή στην καινοτομία και στις ε, ε, επιχειρήσεις που βρίσκονται σε διαδικασία μεταμόρφωσης. Χρειαζόμαστε δηλαδή ε, μια καινοτομία η οποία θα είναι πρωτοπόρα. Το δεύτερο μήνυμα είναι, είναι ένα αίσθημα που το είχα και νωρίτερα, ε, αλλά δεν μπορούσα να το αποδείξω, ότι τα συστήματα υποστήριξης και επιδότησης είναι πάρα πολύ περίπλοκα, γραφειοκρατικά και πολύ περιοριστικά. Αυτό προκύπτει σαφώς από τις απαντήσεις που λάβαμε. Και τρίτον, ότι τα χρήματα από μόνα τους δεν αποτελούν πανάκια. Και τις απαντήσεις αυτές τις έδωσαν άνθρωποι που έχουν ιδρύσει νεοπαγείς ε, εταιρείες, οι οποίοι μου έχουν πει ότι προφανώς χρήματα χρειάζονται, αλλά δεν επαρκούν από μόνα τους. Χρειάζεται να γίνονται και άλλα πράγματα. Χρειαζόμαστε εκπαιδευτές, χρειαζόμαστε καθοδηγητές, ανθρώπους που θα γνωρίζουν πώς θα μας καθοδηγήσουν στο μέλλον. Τους επόμενους μήνες λοιπόν θα αρχίσουμε να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Οπότε θα ήθελα να διατρέξω αυτές τις αλλαγές που σκοπεύουμε να κάνουμε. Πρώτον, πρέπει να προσαρμόσουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε προκειμένου να άρουμε τους περιορισμούς που υπάρχουν. Και σκοπός μας είναι να υπάρξει μια προσέγγιση από τα κάτω προς τα πάνω. Στις ε, μικρομεσίες επιχειρήσεις υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία στη μεταποίηση ή στην ανοτεχνολογία. Εμείς θέλουμε λοιπόν να κάνουμε κάτι που θα έχει μια προσέγγιση από τα κάτω προς τα πάνω. Αυτό είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο που θέλω να συζητήσω μαζί σας. Επίσης, θα θέλαμε επίσης, να αξιοποιήσουμε καλύτερα την γκάμα χρηματοδοτικών εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας και δεύτερον πρέπει να ξαναεξετάσουμε την, ε, τον τρόπο με τον οποίο ε, επιλέγονται τα ε, χρηματοδοτούμενα, χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Κανείς δεν πρόκειται να επενδύσει σε κάποιο project αν δεν ε, γνωρίσει πρώτα τους ανθρώπους που θα ήθελαν να υλοποιήσουν το συγκεκριμένο project. Και τρίτον, ε, δαπανούμε αρκετό χρόνο στην επιλογή των, ε, των προγραμμάτων αλλά δεν δίνουμε αρκετό χρόνο στην, στη συνέχεια που δίνεται και στην παρακολούθηση. Επίσης, πρέπει να αυξήσουμε την ορατότητα των καινοτόμων εταιριών. Επίσης, χρειαζόμαστε εμπειρογνωμοσύνη από ανθρώπους που έχουν δοκιμαστεί στην αγορά, που έχουν ιδρύσει επιχειρήσεις, άλλοτε με επιτυχία, άλλοτε και όχι. Οπότε, αυτές είναι οι αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε. Διακόψτε με, Πρόεδρε, αν ε, υπερβώ το χρόνο μου. Απλά θα ήθελα να σας πω και για το European Science Cloud για τον έφος των επιστημών της Ευρώπης. Αυτό ε, να σας πω δύο λόγια. Γνωρίζετε ότι ε, έχετε ήδη αποφασίσει να με βοηθήσετε στην επίτευξη αυτού του στόχου, να αποκτήσει η επιστήμη μας έναν πιο ανοιχτό χαρακτήρα, γιατί αυτό είναι πραγματικά η ουσία αυτής της πρωτοβουλίας μας και χαίρομαι πολύ που αποφασίσατε να με βοηθήσετε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο της ανοιχτής επιστήμης μέσω έκθεσης της Επιτροπής Ήτρε του κυρίου Σαφχάουζερ που ήταν εισηγητής. Θα ήθελα λοιπόν να τον ευχαριστήσω και προσωπικά. Συγγνώμη και αν προφέρω λάθος το όνομά του. Η Κομισιόν λοιπόν εξέδωσε αυτήν την ανακοίνωση για το European Science Cloud στις 19 Απριλίου του 2016 και παρουσιάσαμε και μια δέσμη μέτρων. Όταν λοιπόν μιλάμε για το European Science Cloud στην πραγματικότητα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να βοηθήσουμε τους επιστήμονες να μπορούν να επαναχρησιμοποιούν τα δεδομένα, τα επιστημονικά δεδομένα που έχουν στα χέρια τους και πώς μπορούν να διαμορφώσουν με βάση αυτά τα δεδομένα το μέλλον. Έχουμε πλέον μια πλειάδα δεδομένων στα χέρια μας και πρέπει πλέον να δούμε πώς σε ένα εντελώς διαφορετικό πλέον περιβάλλον να επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα, όχι πια όπως παλιά που δεν είχαμε δεδομένα, αλλά πλέον πώς θα επιλέγουμε τα σωστά δεδομένα και πώς θα τα αναλύουμε. Αυτό λοιπόν είναι ε, ο σκοπός του European Science Cloud. Δεν είναι μόνο δηλαδή η επιστήμη αυτή καθεαυτή, αλλά και οι υπηρεσίες Είχαμε άλλωστε και μια ομάδα υψηλού επίπεδου που, μας, που μελέτησε το θέμα και μας έδωσε κάποιες ε, ε, συστάσεις και όσον αφορά τη διακυβέρνηση και ε, γι' αυτό λοιπόν ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τη συζήτηση κάποια στοιχεία. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα ε, σημαντικά στοιχεία και όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν τα οποία ε, ε, σχετίζονται με τον ορίζοντα 2020 θα είναι by default ανοιχτά για το 2017. Συμφωνώ επίσης ότι το Συμβούλιο αποφάσισε για την δημοσιοποίηση των στοιχείων και αυτό είναι ιστορική σημασία ε, στοιχείο ε, και με τον τρόπο αυτό τα στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα στην Ευρώπη θα είναι διαθέσιμα και σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήθελα επίσης να καλωσορίσω εδώ ε, και την έκθεση, την πρωτοβουλία μάλλον και απόφαση της Επιτροπής σας Ήτρε να εκπονήσει γνωμοδότηση της κυρίας Καμπεσόν σχετικά με τα θέματα αυτά. Αυτή η ε, έκθεση θα αποτελέσει προστιθέμενη αξία για μένα αυτή, δηλαδή της αξιολόγησης του ορίζοντα 2020. Αυτά ήθελα να σας πω, ελπίζω να μην μακρηγόρησα υπερβολικά. Θα, θα επανέλθω και στις απαντήσεις μου σε ορισμένα από τα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε ε, Επίτροπε για τις εισαγωγικές σας παρατηρήσεις επί τριών πολύ σημαντικών ε, θεμάτων τα οποία μας είναι ιδιαίτερος προσφυλή και ε, τα θεωρούμε ιδιαίτερος σημαντικά. Τώρα, πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Κάρινο εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Ο κύριος Μπάλεαν. Ευχαριστώ που ήρθατε στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας. Η ερώτησή μου αφορά αυτά που είπατε. Διαβλέπουμε τώρα την ε, σημασία ε, των όσων λέτε. Αλλά ξέρετε, ε, εδώ μιλάμε λίγο με σχετικούς αριθμούς ε, σχετικά με το Συμβούλιο καινοτομία. Ε, αλλά αυτό μου θυμίζει λίγο τον χρόνο κοίηση. Στου ελέφαντε μπορεί να είναι 10 μήνε, σε άλλα είδη μπορεί να είναι πολύ περισσότερο, σε άλλα λιγότερο. Νομίζω ότι ε, θα πρέπει να καθοριστούν πιλωτικά προγράμματα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, χρονικά δηλαδή. Επίσης, αναφέρεστε για συζητήσεις που έχουν γίνει όσον αφορά την πληροφορία και την, ε, την τεχνολογία, αλλά εγώ ε, βλέπω ότι ε, άλλοι ασχολούνται με την καινοτομία, άλλος επίτροπος ασχολείται ε, με την τεχνολογία. Ε, έχουμε τέσσερα δις προϋπολογισμό για τέτοιου είδους προγράμματα καινοτομία, τα οποία όμως μοιράζονται σε διάφορες γενικές διευθύνσεις το EIC ενδεχομένως θα πρέπει κάπως να δομήσει καλύτερα ε, τις ε, διάφορες διαδικασίες και τα διάφορα προγράμματα. Ε, θα πρέπει να ξεπεράσουμε κάποια προγράμματα. γιατί ο καθένας δεν θα πρέπει να, ενδιαφέρεται πού θα πρέπει να ενδιαφέρεται το πρόγραμμά μου, στα smart cities, στο, στα προγράμματα IT, δεν ξέρω πώς θα τα συντονίσετε αυτά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ε, στις δύο τελευταίες θητείες δεν είδαμε ποτέ τόσο μεγάλο καταγερματισμό για την καινοτομία όσο βλέπουμε τώρα. Δεύτερον, αναφερθήκατε ε, στην προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, bottom-up. Αυτό είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιδέα θα πρέπει να αφορά όλα τα στοιχεία τα οποία λαμβάνεται ε, από τους εμπλεκομένους ε, και το, η προσέγγιση αυτή bottom-up από κάτω προς τα πάνω είναι φιλικότερη προς τους ε, ε, επιχειρηματίες, ε, προς τους ε, εμπλεκόμενους, αλλά θα πρέπει να έχουν και αυτοί κάποιο χρονοδιάγραμμα. Και για να μπορέσουμε να διευρύνουμε το πρόγραμμα FTI θα πρέπει να έχουμε καλές καλή διάδραση ας πούμε με, του, με τους ε, εμπλεκόμενους. Όσον αφορά τώρα το Open Science Cloud, ε, υπάρχουν κάποιες υποβόσκουσες ε, τριβές μεταξύ διαφορετικών μονάδων και γενικών διευθύνσεων και αναρωτιόμαστε, ναι, το cloud μπορεί να είναι αρτητή, αλλά υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία ενδεχομένως αποτελέσουν ε, σημεία αμφισβήτησης από άλλες γενικές διευθύνσεις. Αναρωτιέμαι λοιπόν πού βρίσκεται η κόκκινη γραμμή ή μάλλον ποιο είναι αυτό, ποια είναι η κόκκινη γραμμή που θα πρέπει να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Εξ των Σοσιαλιστών, ο κύριος Νίκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ αλλά και για την διαρκή σας διαθεσιμότητα για διάλογο. Ε, Open Science Cloud, Αριστεία και το ενιαετές πρόγραμμα πλαίσιο με απασχολούν. Η πρωτοβουλία σας ε, για τον έφος ε, είναι, μας ικανοποιεί. Ανοιχτό λοιπόν νέφος ε, το οποίο ε, θα βοηθήσει 1,7 εκατομμύρια ερευνητές και περίπου 70 εκατομμύρια εμπορευόμενους ε, οι οποίοι ενδιαφέρονται ιδιαίτερος για αυτήν την εξέλιξη των δεδομένων. Το 2016 ε, μέσω της πρώτης έκθεσης ε, ταυτοποιήθηκαν ε, τα πρώτα προβλήματα, η έλλειψη δηλαδή ομοιογένειας της αγοράς, η έλλειψη πραγματογνωμόνων για το θέμα. Εγώ ρωτώ ποιες είναι οι πρακτικές ημερομηνίες, τα πρακτικά στοιχεία για την υλοποίηση. Δεύτερον, όσον αφορά την παραγωγή γνώσης, πρέπει να σας πω ότι ενώ έχουμε καλή έρευνα ε, δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε το αποτέλεσμα της έρευνας ε, και εν πάση περιπτώσει αυτό είναι σημαντικό. Εξίσου σημαντική είναι και η δυνατότητα πρόσβασης ε, στην χρηματοδότηση των, επιστήμων, επιστημόνων, ερευνητών κλπ. Τρίτον, όσον αφορά ε, το ένα το ε, πλαίσιο, πώς, ε, πρόγραμμα πλαίσιο, πώς η Κομισιόν προτίθεται να αντιμετωπίσει αυτό το πλαίσιο. Τα κράτη-μέλη πρέπει να εμπλακούν, αλλά και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμπλακεί επίσης. Θα θέλαμε να ξέρουμε ε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας ε, για το ένα το ε, πρόγραμμα πλαίσιο από το 21 μέχρι το ε, 27. Είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ και βεβαίως χαιρόμαστε που είσαστε εδώ και μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφε. ECR Κύριε Επίτροπε, ο κύριος Χένκελ. Μέχρι το 2020 η Βρετανία προφανώς θα είχε εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αλλά αποτελεί έναν από τους ε, πιο σημαντικούς ε, καθαρούς συνεισφέροντες ε, επομένως, έχετε κάποια ιδέα ε, του ποσοστού του προϋπολογισμού του Ηνωμένου Βασιλείου για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020. Δεύτερον, το Ηνωμένο Βασίλειο εμπλέκεται στον ε, ορίζοντα 2020 ως καθαρός συνδρομητής. Προτίθεστε να διατηρήσετε μέσο και μακροπρόθεσμα ε, τα αρχικά προβλεπόμενα όρια προπολογισμού για το πρόγραμμα ορίζοντας 2020. Εάν τώρα προτίθεστε να κρατήσετε τα ίδια όρια και τους ίδιους προϋπολογισμούς, από πού νομίζετε ότι θα ε, προέλθουν τα χρήματα που θα λείψουν, θα χρησιμοποιήσετε τον υφιστάμενο προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε για τις πολύ συγκεκριμένες και σύντομες ερωτήσεις σας. Εξ ονόματος της Άλντε η κυρία Κάλλας, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση η οποία σχετίζεται και με αυτά που είπε ο συνάδελφος από το ΕΛΚ ε, σχετικά με το Συμβούλιο Καινοτομίας. Στην Ευρώπη λοιπόν έχουμε πολλά καλά πράγματα, καλή βιομηχανία, καλή έρευνα, αλλά ε, λείπουν οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων τομέων. Αναρωτιέμαι εάν το Συμβούλιο Καινοτομία μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα. Έχουμε ε, το, θέμα με τα ΚΙΚΣ, έχουμε τα, θέματα με την πληροφορία ε, και την ε, τεχνολογία. Όλη αυτή η γνώση λοιπόν για την καινοτομία θα πρέπει κάπως να συνδυαστεί με τους άλλους σχετικούς τομείς θα το αντιμετωπίσει αυτό το Συμβούλιο Καινοτομία και κάτι άλλο σχετικό. Ε, ε Συμβούλιο Έρευνας υπάρχει. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολύ καλή έρευνα στην Ευρώπη, αλλά δεν καταλήγει σε καινοτομία στην Ευρώπη. Καταλήγει σε καινοτομία σε άλλες χώρες. Εάν δημιουργήσουμε τώρα ένα ξεχωριστό σώμα για την καινοτομία, στην ουσία θα υπογραμμίσουμε ακόμα περισσότερο αυτήν την διάσταση ε, που υπάρχει, αυτό το κενό που υπάρχει. Ε, το θέμα είναι πώς μπορεί να κινηθεί το Συμβούλιο Έρευνας και Καιροτομίας έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Επίτροπε. Και εγώ θέλω να μια ερώτηση σχετικά με το θέμα το πρώτο, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καινοτομία. Προβληματίζομαι λίγο. Έχετε ήδη κάνει μια σχετική πρόταση από όσο ξέρω. Θα ήθελα όμως εγώ να σας μιλήσω για την συμμετοχή ε, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο καινοτομίας της Ευρώπης, γιατί εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ε, δηλαδή, η κύρια ραχοκοκαλιά, ας το πούμε, παραγωγική ραχοκοκαλιά της Ευρώπης ε, αποτελείται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, πώς είναι δυνατόν ε, αυτές οι μικρές εταιρείες να συμμετάσχουν στην καινοτομία. Τώρα ε, την καινοτομία την παράγουν κυρίως ε, οι μεγάλες εταιρείες, ε, οι πολυεθνικές. Υπάρχει όμως τεράστια, τεράστιο δυναμικό καινοτομίας. Πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό, πώς μπορούμε να ελέγξουμε τη διαδικασία μετακίνησης χρημάτων προς αυτές τις πολυεθνικές εταιρείες έτσι ώστε να σταματήσει αν γίνεται και να κινηθούν χρήματα και προς τις μικρότερες. Δεύτερον, μία ερώτηση. Ποια θα είναι η διασύνδεση ανάμεσα στο Συμβούλιο Καινοτομίας και το ονομαζόμενο ε, σχέδιο Juncker, δηλαδή το πρόγραμμα στρατηγικών επενδύσεων. Θα, η διασύνδεση θα είναι μέσω του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Φαντάζομαι ότι το Ινστιτούτο αυτό δεν έδωσε εν τέλει τα προβλεπόμενα αποτελέσματα. Ε, ξέρω ότι δεν θέλετε να δημιουργήσετε νέους οργανισμούς, αλλά παρόλα αυτά πώς ε, θα γίνει η διάρθρωση και η διασύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα διαφορετικά εργαλεία, γιατί η διασύνδεση δεν υπάρχει για την ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπορέλη, η FDD. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την παρουσία του. Τον ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων. Υπογραμμίσατε την ε, δυσκολία που έχουν οι επιχειρήσεις στην χρήση αυτών των ε, εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς για να βοηθήσουν την καινοτομία. Ορθώς επίσης υπογραμμίσατε το γεγονός ότι αυτά τα εργαλεία δεν είναι τόσο γνωστά όσο θα έπρεπε και επομένως θα πρέπει να αυξήσουμε τις προσπαθειές μας κατά αυτή την έννοια προκύπτει όμως και ένα άλλο ερώτημα. Υπάρχουν πολλές ε, εταιρείε οι οποίες γνωρίζουν τα εργαλεία αυτά συμμετέχουν θεωρείται σωστό και καινοτόμο το πρόγραμμά τους, αλλά μετά δεν λαμβάνουν την απαραίτητη χρηματοδότηση, διότι ε, δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή. Ερώτηση λοιπόν, είναι δυνατόν στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, να ε, υπάρχει δυνατότητα να καλυφθούν ε, τέτοια πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κινητοποιηθούν τουλάχιστον ένα μισό δις ευρώ έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν αυτές οι μικρές εταιρείες οι οποίες είναι έτοιμες για την καινοτομία αλλά δεν λαμβάνουν τελικά την χρηματοδότηση. Χρειάζεται αυτή την μικρή όθηση η ε, ε, καινοτομία μέσω των μικρών μεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Το χρειάζεται και η Ευρώπη αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα και εγώ να σας χαρώ για την ε, νίκη της Πορτοκαλίας. Ε, και και τις δύο πλευρές εγώ το σκεφτόμουν, ε, όπως και να έχει όμως, είτε η Γαλλία κέρδισε την Πορτοκαλία εγώ χαρούμενος θα ήμουν, είμαι και σήμερα λοιπόν. Έχω πολλές ερωτήσεις κύριε Επιτροπέ. Η πρώτη αφορά το περιβάλλον. Κατανοώ ότι δική σας ανησυχία αφορά περισσότερο τις υπηρεσίες και τη διακυβέρνηση ε, σε ό,τι αφορά την επιστημονική κοινότητα. Δεν αφορά δηλαδή απευθεία ε, την τεχνολογία. Για το περιβάλλον, λοιπόν, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε το θέμα του υπολογιστικού νέφους ε, χωρίς να δούμε το... την αποθήκευση δεδομένων δηλαδή, γιατί το νέφος δεν σημαίνει κάτι από μόνο του. Θα μπορούσαμε λοιπόν να σκεφτούμε αυτό το ζήτημα χωρίς να εξετάσουμε ε, τις δημόσιες ελευθερίες ε, και την κυριότητα αυτών των ε, δεδομένων. Μπορούμε λοιπόν να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα χωρίς να θέσουμε το ζήτημα ποιος παίρνει αυτά τα δεδομένα. Έχει το δικαίωμα να τα αξιοποιήσει και υπάρχει και από πλευράς πολίτη αποδοχή για την χρήση και αξιοποίηση των δεδομένων. Γενικά, ας πούμε, βλέπουμε ότι παίρνουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να θεωρούμε φυσιολογικό και πρέπει εμεί να δηλώσουμε την αντίθεσή μας, ας πούμε, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Ή γενικά είναι φυσιολογικό ε, την κυριότητα αυτών των δεδομένων την έχει αυτός που τα παράγει είναι ένα θέμα ουσίας. Δεν μπορούμε να προωθήσουμε το ζήτημα του νέφους χωρίς να εξετάσουμε αυτό το θέμα. Δεύτερον, είπατε ότι δεν εξετάζουμε την ε, πλευρά της τεχνολογίας που παίρνουμε κατευθείαν στις υπηρεσίες. Όμως για μας, τι συμβαίνει με τα software, τα hardware, με αυτά που έχουμε εδώ στην Ευρώπη και το θέμα και πάλι της κυριαρχίας. Ξέρετε πόσο σημαντικά είναι τα PIN και είστε τραπεζικό είστε, αρκεί να βάλει κανεί μερικά τέτοια πιν σε ένα σύστημα τραπεζικών συναλλαγών και ε, ξαφνικά κάποιο μπορεί να γνωρίζει ε, όλες τις τραπεζικές συναλλαγές. Εγώ προέρχομαι από τον χώρο του στρατού και σε ορισμένε περιπτώσει δεν ήμασταν σίγουροι αν ήμασταν ε, σε αντίθεση με τον ΝΑΤΟ όταν υπήρχε ας πούμε ε, μία κίνηση ενός Ραφάλ. Έχουμε λοιπόν ένα τεχνολογικό στοιχείο το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και στο software και στο hardware. Γιατί να έχει κάνει στο λογισμικό χωρίς να έχει το hardware δεν έχει νόημα. Πρέπει λοιπόν να τεθεί και αυτό το ζήτημα. Και εσείς δεν το πιστεύετε αυτό. Τώρα, για να πούμε στο θέμα, αυτό καθ' αυτό, δηλαδή τις υπηρεσίες που αναφέρατε είναι ένα πρώτο ερώτημα που πρέπει να λύσουμε. Μήπως η ανοιχτή ανταλλαγή δεδομένων οδηγεί στην καινοτομία. Ισχύει αυτό ή όχι. Πρέπει να θέσουμε αυτό το ζήτημα. Εγώ έχω εμπειρία στο τομέα της καινοτομίας, ιδίω ό,τι αφορά την ασφάλεια, την αμυντική, αλλά και στους δορυφόρους. Από την ανοιχτή ανταλλαγή των δεδομένων φτάνουμε. Γιατί τελικά η χώρα μου είναι σχεδόν η μοναδική που κατέχει αυτές τις τεχνολογίες στην Ευρώπη. Από αυτό το είδος ανταλλαγών δεδομένων φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Να είμαστε από τις ηγέτητες δυνάμεις ε, στους δορυφόρους, ε, στην αεροπλοεία. Υπερθυμίζω για παράδειγμα ότι ένας υπολογιστής Ραφάλ ε, κάνει μεγαλύτερη δουλειά από ότι το Dispatching Center ε, στη Γαλλία. Έχει μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ. Επομένως, από τη δική μου εμπειρία για την καινοτομία, βλέπουμε ότι έχουν περισσότερο κλειστές ερευνητικές κοινότητες, εξειδικευμένες, και η καθεμία έχει αναλάβει ένα μικρό τμήμα. Για παράδειγμα, στην Airbus, ο Διευθυντής Ερευνών της Airbus, τον οποίο γνωρίζω, δείχνει ότι είναι απολύτως αδύνατον να λειτουργήσει από κοινού η γερμανική και γαλλική ερευνητική κοινότητα. Δεν θα οδηγούσε αυτό πουθενά. Και καλύτερο θα ήταν να γίνει εξειδίκευση, οι ε, Γάλλοι κάνουν περισσότερη έρευνα, οι Γερμανοί marketing και βιομηχανοποίηση. Και αν θέλουμε να τους βάλουμε όλους σε όλα και με διαφορετικές κουλτούρες δεν έχει κανένα νόημα στην έρευνα. Μετά κάτι αεροσκάφη, ας πούμε, που απασχόλησαν και τα ευρωπαϊκά ερευνητικά πρόγραμμα. Δεν κάναμε όλοι τα πάντα, τα μοιράσαμε. Μήπως θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα. Μετά τίθεται το ζήτημα της διακυβέρνησης. Και εδώ έχω κάτι να αναφέρω. Είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν με τις υπηρεσίες σας για να μπορέσουμε και εμείς ε, να συμβάλλουμε με θετικό τρόπο, χωρίς όμως να ξεχνούμε και το περιβάλλον. Ε, παρότι κατανοώ ότι δεν είναι το κύριο ζήτημα εδώ, παραμένει όμως σημαντικό. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει μια θετική συμβολή. Σας ευχαριστώ κύριε Πίτροπε και ευχαριστώ και σας κύριε Πρόεδρε που ε, με αφήσατε λίγο να μακρηγορήσω. Ευχαριστώ. να δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει. Στον πρώτο γύρο ερωτήσεων έχουμε ακόμα 12-13 συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο στο δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ξεκινώ τον κύριο Έλερ και την κυρία Κάλλας. Ο κύριος Έλερ μίλησε για την κοίηση. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή μεταφορά. Και να σας πω για το χρονοδιάγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομία και αυτό απευθύνεται και στην κυρία Κάλλας. Ξεχνά, ξεχάστε τον όρο Συμβούλιο, σχεδόν μπορώ να πω. Εδώ δεν θέλουμε να συστήσουμε ένα νέο φορέα, δεν θέλουμε να έρθουμε σε αντίθεση με τους ε, ήδη φυστάμενους θεσμούς. Θέλω λοιπόν να σας περιθμίσω ορισμένα πολύ συγκεκριμένα πράγματα που θέλουμε να κάνουμε και μπορείτε μετά να πείτε κι εσείς τι είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καιροτομίας. Είναι αυτά τα, τα, οι δέκα εργασίες που θέλουμε να αναλάβουμε, τα δέκα καθήκοντα, χωρίς όμως να αλλάξει καθόλου το νομικό πλαίσιο. Χρειαζόμαστε λοιπόν μία ομάδα συμβούλων στην καινοτομία. Όπως και στην έρευνα έχουμε 7 τέτοιους ε, επικεφαλείς συμβούλους ερευνών. Έχουμε και εδώ λοιπόν συμβούλους καινοτομία, ανθρώπους που έχουν ανοίξει επιχειρήσεις και ούτω καθεξής. Μετά, θέλαμε να αναθεωρήσουμε το πρόγραμμα εργασιών 2000, του ορίζοντα 2020 με μια απλή εκπροσώπηση και παρουσίαση των ε, εργαλείων για να ξέρουν όλοι πού να πάνε, με απλές διαδικασίες, τα βραβεία και το καθεξής, γιατί είναι πολύ περίπλοκο. Αυτό μου λένε πολλοί νέοι επιχειρηματίες. Μετά, οι μικροπιστές επιχειρήσεις, να τις καλούμε με μια bottom-up διαδικασία, με συνεχείς εκκλήσεις, ε, προσκλήσεις ε, υποβολής ενδιαφέροντος. Θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε αυτή την ε, βασική ιδέα. Η κυρία Κάλλας μίλησε για το, το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Συμβούλιο. Το μόνο που μου έχουν δώσει ως σχόλιο για το τι πρέπει να κάνουμε παραπάνω δεν είναι να κάνουμε περισσότερα, είναι να έχουμε αυτή την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω. Μετά, κριτήρια αξιολόγηση. Πώς μπορούμε να τα ενισχύσουμε για να επικεντρωθούμε ε, στις καινοτομίε που διαμορφώνουν αγορές αυτές οι καινοτομίες που αναφέραμε προηγουμένως. Και μετά πρέπει να αναθεωρήσουμε και να επιταχύνουμε τη δικασία αξιολόγηση με ε, συνεντεύξεις, με ομάδες, με ταχύτερα αποτελέσματα. Σε αυτά τα πράγματα και εδώ. Μετά, πρόσβαση στους ε, αυτούς τους mentors, ε, του συμβούλους καθοδήγησης, ας πούμε. Κάποιες φορές δεν ξέρουμε, μετά την στήριξη που δίνουμε σε επιχειρήσεις, δεν ξέρουμε τι απογίνονται αυτές. Μετά να δούμε νέα μέσα ε, κλιμάκωσης ε, των ε, επιχειρήσεων. Scale up. Να το δούμε λοιπόν, κατά πόσο υπάρχουν και εκεί κάποιες ε, θετικές προτάσεις. Δεδομένα και στοιχεία σε πραγματικό χρόνο, για να έχουμε περισσότερα δεδομένα και ε, εταιρικέ σχέσει με υφιστάμενες πρωτοβουλίες και η πύλη ορίζοντα 2020. Αυτά είναι τα 10 καθήκοντα που έχουμε αναλάβει. Και για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητα, όταν μιλάμε, αυτό εννοούμε. Αυτό θέλουμε να κάνουμε τώρα. Και γι' αυτό θέλω τη στήριξή σα. Είναι καλό αυτό που λέτε, να στηρίξουμε την ε, βιομηχανία, να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε πιο άμεση επαφή. Ο κύριος Έλλερ ε, έθιξε το σημαντικό ζήτημα των, της διάρθρωσης μεταξύ των επιμέρους γενικών διευθύνσεων. Εγώ είμαι υπέρμαχος της συνεργασίας μεταξύ των γενικών διευθύνσεων. Βρίσκομαι λοιπόν σε άμεση επαφή με το EIT, με τον συνάδελφό μου Ντομπρόφσκης, όμως ε, κατανοώ και αυτό που λέτε. Πρέπει κάπως να αρθούν ε, αυτά τα στεγανά. Δεν μπορούμε να κατακριτήσουμε σε τέτοιο βαθμό τη δουλειά μας. Για το fast track για την καινοτομία, κύριε Έλλερ, νομίζω ότι είναι καλή ιδέα και καλό παράδειγμα ε, σαν πιλωτικό έργο ουσιαστικά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το πάνω από χίλιες τέτοιες προτάσεις, 62 προγράμματα έχουν χρηματοδοτηθεί, σημαντικά ποσά έχουν ταπανηθεί. Μόνο και μόνο για αυτό το μέσο. Είναι λοιπόν μεγάλη επιτυχία. Ο κύριος Νίκα στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ε, με ρωτήσατε για το ερευνητικό νέφος. Έχουμε λάβει αυτή την έκθεση από τις ε, ομάδες εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου. Αυτά τα milestones, λοιπόν, οι βασικές ημερομηνίε είναι την Άνοιξη του 2017 θα έχουμε οδικό χάρτη για τη διακυβέρνηση και χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Νέφους που θα βασίζεται κυρίως ε, σε αυτές τις συζητήσεις των εμπειρογνωμόνων. Η ομάδα υψηλού επίπεδου που ε, δημοσιοποίησε αυτή την έρευνα μα έδωσε καλέ προτάσει ό,τι αφορά την πολιτική, τη δικυβέρνηση και την υλοποίηση. Θα τα μελετήσουμε λοιπόν. Όλα τα δεδομένα που θα προκύπτουν από το ορίζοντα 2020 by default θα είναι ανοιχτά και διαθέσιμα από το 2017 και θα επανέλθω στην παρατήρηση ε, του εισηγητή για τα δεδομένα για να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τα χρήματα των φορολογουμένων και να δώσουμε κίνητρα για την καινοτομία. Αυτό ε, θα επιτευχθεί και με μελλοντικά προγράμματα στο ΡΙΖΟ 2020. Τα τελευταία τρία χρόνια του 2020 θα τα βελτιώσουμε περαιτέρω για να τα ε, συντονίσουμε με άλλα ε, καταγραμματισμένα μέσα που έχουμε αυτή τη στιγμή για να δούμε πώς μπορούμε πιο φθηνά και πιο αποτελεσματικά να εργαστούμε προς όφελος του Ευρωπαίου πολίτη. Έχουμε και τη διαρκή σας στήριξη και σας ευχαριστώ. Μετά, με ρωτήσατε για τις ε, μελλοντικές προθεσμίες για το πρόγραμμα πλαίσιο 9. Από το, μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2016 θα έχουμε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση για την ενδιάμεση αξιολόγηση. Μετά το Δεκέμβριο θα αρχίσει η εναρτήρια συνάντηση ε, της ομάδας ψηλού επίπεδου. Τον Γενάρη του 2017 έχουμε την κοινή αυτή εκδήλωση των ενδιαφερμένων μερών. Μετά μέχρι τον Οκτώβριο του 2017 θα κινηθούμε γύρω στο Μάη θα έχουμε τη δημοσίευση του Staff Working Document, μετά έκθεση στην ομάδα ψηλοεπιπέδου, μετά ε, τα σχόλια του Κοινοβουλίου και μέχρι τον Οκτώβριο του 2017 θα έχουμε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενδιάμεση αξιολόγηση του Horizon 2020 και τις μελλοντικές προβλέψεις για το ένατο πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτά είναι τα βήματα που με ρωτήσατε και ήθελα να σας ε, ενημερώσω. Μετά η ερώτηση του κυρίου Χέγκελ. Με ρωτήσατε λοιπόν για το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρώτα απ' όλα. Γνωρίζουν όλοι αυτά που έχουμε κάνει με το Ηνωμένο Βασίλειο και όσοι με γνωρίζουν γνωρίζουν πόσο έχω στεναχωρηθεί για την εξέλιξη αυτή. Αυτή τη στιγμή όμως η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του Ηνωμένου Βασιλείου. Οπότε εγώ δεν μπορώ να σας πω και πολλά πράγματα. Τα πράγματα έχουν ως έχουν αυτή τη στιγμή. Δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχουμε ενημερωθεί για κάποια αλλαγή, θεσμικά τουλάχιστον. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε όπως έχουμε πει ότι θα το κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε νέε συζητήσει σε διάφορου τομεί. Γιατί αυτό νομίζω ότι θα έβλαπτε την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή η μπάλα, το μπαλάκι βρίσκεται στην πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αλλά από εκεί και πέρα θα δούμε και πώ θα κινηθούμε. Γνωρίζω ότι αυτά τα, αυτά τα ερωτήματα απασχολούν όλου μα και τα δεχόμαστε κι εμείς ε, διαρκώς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να, παρά μόνο να σας πω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να είναι μέλος της Ένωσης και ότι προφανώς ε, ε, η κατάσταση πράγματι, κύριε Χένκελ, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μετά, είχα ένα ερώτημα από την... Ε, συμπατριώτησά μου, τη Μαρίζα Ποτήσου, οπότε θα μιλήσω λίγο πορτοκαλικά με την ευκαιρία και μετά θα επανέλθω στα ε, αγγλικά. Σας ευχαριστώ πολύ ε, κυρία Βουλευτά για τις ε, πολύ σωστές ερωτήσεις σας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τεχνολογία, ε, Καινοτομίας προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία θίξατε. Ας πούμε ποια είναι η θέση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πώς μπορούμε να αποφύγουμε τα προβλήματα, πώς ε, μπορούμε να ενεργήσουμε έτσι ώστε να μην είναι πάντα οι ίδιοι οι οποίοι ε, ε, εντάσσονται στα προγράμματα. Γνωρίζουμε ότι συχνά τα τα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με τον ορίζοντα 2020 δεν γίνονται γνωστά στο ευρύ κοινό. Εμείς θέλουμε ακριβώς να προσεγγίσουμε τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Θέλουμε αυτή την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω, γιατί γνωρίζουμε ότι η πλοήγηση αυτών των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων είναι τέτοια που δεν τολμούν να ε, παρέμβουν ε, σε αυτά τα προγράμματα ε, της καινοτομίας. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εταιρείε. Θα μπορέσουμε επίσης να δούμε ποια είναι τα ασθενή και ισχυρά σημεία του προγράμματος Επίσης αναφερθήκατε, με ρωτήσατε ποια είναι η διασύνδεση ανάμεσα στο σχέδιο Juncker και την τεχνολογία. Κοιτάξτε, είναι λίγο σαν σούπα. Έχετε όλα τα στοιχεία, τα, όλα τα συστατικά, τα οποία τα έχετε βάλει στον πάγκο της κουζίνας, ε, ε, το σχέδιο Juncker, τα άλλα προγράμματα, το Συμβούλιο ε, και το Συμβούλιο της Καινοτομίας είναι η κατσαρόλα μέσα στην οποία θα μπουν όλα τα στοιχεία για να φτιαχτεί η ωραία η σούπα. Δηλαδή αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι ένα μείγμα ε, από τα διάφορα στοιχεία τα οποία ε, θέλουμε να ε, λάβουμε υπόψη μας. Για την χρηματοδότηση. Κύριε Μπορέλη, θα ήθελα να αναφερθώ με την ευκαιρία αυτή σε ένα θέμα το οποίο δεν, για το οποίο δεν μίλησα. Το ζήτημα της αριστείας πρώτον. Πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι συνέργειες μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και νομίζω ότι η χώρα σας είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει και να προωθήσει κανείς την αριστεία. Η Ιταλία έχει σημειώσει εκπληκτικές επιτυχίες στον ε, τομέα αυτό. Και δεύτερον, για τα ταμεία, επειδή αναφερθήκατε στα 500 εκατομμύρια, ε, ένας από τους στόχους είναι να από τα ταμεία είναι ότι σήμερα δεν είναι δύσκολο να ιδρύσει κανείς μια εταιρεία στην Ευρώπη. Το, το δύσκολο είναι πώς μπορεί κανείς να κλιμακώσει την ανάπτυξη αυτής της εταιρείας και να, να καταστεί μια μεγάλη εταιρεία. Οπότε έτσι αυτό το θέμα βεβαίως θα ε, εντάσσεται, θα συμπεριλαμβάνεται και στο πακέτο για την ε, κεφαλαία αγορά, την ενιαία κεφαλαία αγορά που προετοιμάζουμε. Μετά, κύριε Ζανλουίκ Σοφχάουζερ. Καλά το λέω. Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω στα γαλλικά. Όσον αφορά την αποθήκευση των δεδομένων, κοιτάξτε εδώ οι Ευρωπαίοι ερευνητές, οι Ευρωπαίοι επιστήμονες μας το ζητούν. Γιατί Πρωτίστως διότι διαπιστώνουν ότι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ικανότητα ε, να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες υπηρεσίες και τεχνολογίες. Ε, δηλαδή μερικές φορές δεν ξέρουν πού να αποθηκεύσουν τις ε, πληροφορίες τους. Συχνά στρέφονται προς την Κίνα ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να αναπτύξουμε αυτή την ικανότητα για τους ερευνητές έτσι ώστε αυτά τα στοιχεία να μπορούν να μείνουν στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για την ε, ερώτησή σας, γιατί ίσως δεν ήμουν σαφής ε, στην αρχική μου παρέμβαση. Η τεχνολογία είναι απαραίτητη, αλλά όχι ικανή ε, προϋπόθεση. Θα πρέπει να έχουμε... γιατί καταλαβαίνετε ότι αν έχουμε ακόμα και πολύ προχωρημένη τεχνολογία, εάν δεν υπάρχουν ταυτοχρόνως και όλες οι απαραίτητες υπηρεσίες, ε, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. 90% ε, των δεδομένων στον κόσμο ολόκληρο δημιουργήθηκαν τα δύο τελευταία χρόνια. Για φανταστείτε, είναι τρομερό αυτό. Επομένως θέλουμε να έχουμε τεχνολογία η οποία να είναι ανώτερη από την τεχνολογία που παράγεται σε, άλλες, ε, σε άλλα μέρη του κόσμου και θέλουμε βεβαίως και τις υπηρεσίες που πηγαίνουν παράλληλα. Με ρωτήσατε και κάτι άλλο. Ε, ένα το οποίο αφορά το άνοιγμα και ε, δύο όσον αφορά την διαφοροποίηση. Ε, τώρα έχουμε πλέον πιστεί ότι το άνοιγμα δημιουργεί προστιθέμενη αξία. Εγώ πολύ συχνά αναφερόμουν παλιότερα στο πρόγραμμα του ανθρωπίνου γονιδιώματος που δημιούργησε πάνω από 300.000 θέσεις εργασίας και πάνω από 800 δις. Ήμουν στην Χαϊδελβέργη στο κέντρο της Bioinformatica και ε, αυτή υπολόγισαν ότι το άνοιγμα των δεδομένων μπορεί ε, να οδηγήσει σε αξία 1,2 δις. Αυτό ακριβώς μας δείχνει πώς ε, πλέον πρέπει να μοιραστούμε τα δεδομένα μας, αλλά να προστατέψουμε, να μοιραστούμε τις γνώσεις μας, αλλά να προστατέψουμε τις ιδέες μας. Και συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει να προστατεύουμε τις ιδέες, γιατί οι ιδέες είναι το ε, προϊόν, αλλά δεν μπορούν να προκύψουν νέα προϊόντα εάν δεν υπάρχει ένα μοίρασμα ε, το, και προώθηση των γνώσεων. Τώρα, το δεύτερο σημείο, η διαφοροποίηση. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη. Ε, αυτό κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη, γιατί αυτή η πολυμορφία ε, η πολιτιστική, η θρησκευτική, ε, η, ο τρόπος και η ικανότητα να βλέπουμε τον κόσμο αποτελεί βάση εκ των για την τεχνολογία. Και εγώ αρέσκομαι να λέγω ότι αυτό είναι το καλύτερο στοιχείο που έχουμε εμείς εδώ γιατί έχει άλλωστε μελετηθεί επιστημονικά ότι ακριβώς από εκεί προκύπτει η μεγάλη μας ε, δύναμη όσον αφορά βέβαια αυτά που είπατε για την ε, προστασία των δεδομένων. Είναι όντως ανοιχτά ερωτήματα, δεν έχουμε ακόμα απάντηση σε όλα. Ποιος έχει την κυριότητα αυτών των δεδομένων, θα πρέπει να τα λύσουμε όλα αυτά. Πάντως, εγώ επιμένω ότι το μοίρασμα, η προώθηση των γνώσεων μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Ε, ε, στον επιστημονικό κόσμο εγώ ξέρω ποια είναι η απάντηση και σα την έδωσα. Τώρα στον υπόλοιπο κόσμο και από πολιτική άποψη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. 15 ομιλητέ έχουμε στον κατάλογο, λέει ο Πρόεδρος. Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώ ο κάθε ομιλητή θα έχει στη διάθεσή του ένα λεπτό το ανώτερο. Για να δώσουμε και τη δυνατότητα στον Επίτροπο να απαντήσει βεβαίω τοποθετήσεις ενός λεπτού. Τον κύριο Ζανονάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον κύριο Επίτροπο για την σαφέστατη παρέμβασή του. Ε, θα κάνω μια παρατήρηση που την έχω ξανακάνει και θα ήθελα τώρα να έχω μια πιο σαφή απάντηση. Το Δεκέμβριο του 2014, εννέα κράτη, τα οποία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα μεσογειακά κράτη, Κροατία, Κύπρος, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία ε, υπέβαλαν πρόταση για συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα πρόγραμμα εταιρική σχέσης για την έρευνα ε, και την καινοτομία στην Μεσόγειο, το οποίο φέρει το όνομα Πρίμα. Οι υπηρεσίες της Κομισιόν προχώρησαν σε αξιολογήσεις επιπτώσεων όσον αφορά την πρωτοβουλία αυτή. Ε, παρά την ύψιστη διπλωματική και πολιτική αξία της πρωτοβουλία. η ε, κολλησιεργεί και δεν δίνει την ε, δική της ε, άποψη με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προωθηθεί αυτή η πρωτοβουλία. Θα ήθελα κάποια απάντηση σχετικά με το πού βρίσκονται οι διαβουλεύσεις όσον αφορά το πρίμα και τι προτίθεται να κάνει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Καστίγιο. Βέραμε, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε είναι, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρώτα απ' όλα, ε, ο δικός χάρτης για την ανάπτυξη και διεύρυνση ε, του νέφους. Αυτό είναι κάτι απαραίτητο και απολύτως επίγον. Μας είπατε ε, ότι ίσως από, τον, από το 2017 θα μπορέσουμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και να έχουμε, ε, να έχουμε οδικό χάρτη, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αυτές. Δεύτερον, όπως μόλις είπε ο Ιταλός συνάδελφος, το θέμα αυτό του προγράμματος Πρίμα πρέπει πρέπει από πλευράς της Εκομισιόν να προκύψει νομοθετική ε, πρόταση γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσει να συζητηθεί το θέμα στο Συμβούλιο Ανταγωνισμού του Απριλίου του 2017 και δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει να ενταχθεί μάλλον από το 2018 στο πρόγραμμα πλαίσιο. Επήγει και αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ ε, για το ε, ευρώ, για την αλλά και για την προσέγγιση ε, που έχετε ε, αναλάβει όσον αφορά δηλαδή αυτή την προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω για να βοηθήσετε την τεχνολογία. Ε, όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες δράσεις οι οποίες μας προβληματίζουν. Το κοινό πρόγραμμα έρευνας του ΣΕΣΕΡ δεν θα μπορούσε να δουλέψει πάνω σε τέτοια θέματα. Όλοι οργανώνουν εργαστήρια, workshops και ό,τι θέλετε άλλο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να υπάρχει και ένας κώδικας δεοντολογίας ε, έτσι ώστε να αποφευθούν προβλήματα σαν αυτά που είδαμε πρόσφατα στην αυτοκινητοβιομηχανία και που δυσμενώς ε, ε, επηρεάζουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και πολιτών. Τώρα, ένα άλλο θέμα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη καινοτομίας Πιστεύετε ότι ε, η ιδέα η οποία έχει ξεκινήσει μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένη και να βοηθήσετε κι εσείς σε αυτό. Ο συνάδελφος Μαρτά έχει εγγραφεί στον κατάλογο, αλλά δεν είναι εδώ. Thank you very much, Mr. Ο κύριος Μπόνι. Κύριε Πίτροβε, συγχαρητήρια για την παρουσίασή σας και για τις προσπάθειες που κάνετε προκειμένου να γίνει η ευρωπαϊκή έρευνα πιο καινοτόμα και πιο προσαρμοσμένη ε, στις προκλήσεις. Νομίζω ότι αυτή η έννοια της ανοιχτής ε, καινοτομία και του ανοιχτού επιστημονικού νέφους είναι κρίσιμη σημασία. Αλλά όταν μιλούμε για το επιστημονικό νέφος νομίζω ότι υπάρχουν ακόμη κάποια ανοιχτά ερωτήματα. Πρώτον, πώς μπορεί να αναπτυχθεί η ανάπτυξη να αναπτυχθεί η χρήση δεδομένων με ταυτόχρονο σεβασμό στην προστασία της ιδιωτικότητας όταν μιλούμε για προσωπικά δεδομένα και πώς ο ανοιχτός χαρακτήρας αυτός μπορεί να διευκολύνει την ελεύθερη ροή των δεδομένων στην Ευρώπη στο μέλλον. Δεύτερον, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ε, συνεργασία όλων των χωρών και όλων των επιστημονικών φορέων σε αυτό το επιστημονικό νέφος και τι είδους προώθηση χρειαζόμαστε προκειμένου να διαχείρισουμε αυτές τις πληροφορίες για το ποια θα είναι τα ωφέλη από αυτήν την χρήση του ανοιχτού επιστημονικού νέφους. Και τέλος, ποιες προϋποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται για αυτό το επιστημονικό νέφος. Ε, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε πολύ πιο ανοιχτοί όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία, για παράδειγμα, προκειμένου να μπορούν να ανταλλάσσονται με μεγαλύτερη ευκολία τα επιστημονικά δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπόνι. Κυρία Βερίνκ. Συγγνώμη. Βερίνκ. Συγγνώμη για την προφορά μου. Ε, σας καλωσορίζω κιόλας στην Επιτροπή Ήτρε. Ε, αντικαθιστάτε τον κύριο Ντεμπάκερ. Είστε νέο μέλος της Επιτροπής μας λοιπόν. Είστε το 7ο, 8ο ή 9ο νέο μέλος της Επιτροπής από την έναρξη της κοινοβουλευτικής περίοδου. Έχετε το λόγο. Αγαπητέ κύριε Επιτρόπε, σα ευχαριστώ για την σαφέστατη παρουσίαση. Δύο ερωτήσει. Πολύ συχνά ακούμε ότι πρέπει να βρούμε πλούστερου τρόπου ε, εξασφάλισης Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τι επιχειρήσει και τι μικρομεσαίες. Όμω πολύ συχνά βλέπουμε ότι κάποιες φορές δεν είναι ε, απαραίτητη αυτή η χρηματοδότηση. Εσείς ε, ποια θεωρείτε ότι είναι τα μέτρα για να επιτρέψουμε στις ε, επιχειρήσεις μας να γενοτομήσουν, χωρίς όμως να παραπέ... τους παραπέμπουμε στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Δεύτερον, πολύ συχνά γίνεται λόγος για τις Ηνωμένες Πολιτείες ως πιο καινοτόμα χώρα από ότι οι ευρωπαϊκές χώρες. Οι επιχειρήσεις καινοτομούν ταχύτερα και έτσι μεγαλώνουν κιόλας είπατε ότι πρέπει και εμείς να ε, δώσουμε περισσότερες διευκολύνσεις στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για να παίρνουν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Όμως, πολύ συχνά υπάρχουν και άλλες δυνατότητες, όπως είναι οι ε, επενδύσεις υψηλού ρίσκου στην Ευρώπη. Ε, πώς το χειρίζεστε αυτό. Και τέλος, θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ εσάς και τη χώρα σας για την ε, νίκη σας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πρωτοσφαίρου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, αν κοιτάξουμε εκείνους που έλαβαν χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ορίζοντα 2020, είναι σαφές ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη γεωγραφική κατανομή. Υπάρχουν τα παλιά και τα νέα κράτη-μέλη. Και το ίδιο χάσμα υπάρχει και στο πρόγραμμα Νότερ. Δεν σας ανησυχεί αυτό. Τι μέτρα θα λάβετε για να άρετε αυτόν τον περιορισμό, για να μπορούν και τα... Ε, οι, συμμετω... συμμετέχοντες και από άλλες χώρες να λαμβάνουν χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε πίτροπε. και εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτή την ε, πολύ ωραία νίκη σας ε, στο Euro την Κυριακή. Θα ήθελα κύριε Επίτροπε τώρα να σας ρωτήσω για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελβετίας. Στην δική μου περιφέρεια, στην Ανατολική Γαλλία, ο ερευνητικό κόσμος αλλά και ο επιχειρηματικός ε, είναι βαθιά αλληλένδετοι και συνδέονται μάλλον πολύ βαθιά και με την Ελβετία. Το γνωρίζετε κι εσείς γιατί ήρθατε ε, να εγγενιάσετε το ευρωπαϊκό, ε, την Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιούπολη πριν από μερικές εβδομάδες στο Στρασβούργο. Έχουμε λοιπόν πολύ σημαντικούς δεσμούς ε, με την Ελβετία που είναι πραγματικός εταίρος μας. Έχω λοιπόν το εξής ερώτημα τι γίνεται με την Ελβετία και τη συμμετοχή της στον ορίζοντα 2020. Ξέρω ότι η μερική εταιρική σχέση ε, λύγει ε, στα τέλη του 2016. Πρέπει να υπογραφεί το νέο πρωτόκολλο. Θα γίνει αυτό. Και θα έχει συγκεκριμένες επιπτώσεις σε αυτή τη ε, συμφωνία το Brexit. Ευχαριστώ κυρία Μούντι. Thank you. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να σας συγχαρώ και εγώ για την Κυριακή. Νομίζω ότι ε, θα, θα ήλπιζα μάλλον η ήττα της Αγγλίας να ήταν το χειρότερο που είχε συμβεί αυτό το καλοκαίρι στη χώρα μου, αλλά μάλλον δεν είναι έτσι. Ε, εκπροσωπείται λοιπόν ολόκληρη τη, τη Μεγάλη Βρετανία, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, διάφορα θέματα. Πρώτον, μιλήσατε για την καινοτομία και τις startup εταιρείε. Όσον αφορά την απασχόληση όμως, πραγματικά αυτό το scale-up είναι πολύ σημαντικό, αυτή η κλιμάκωση και η ανάπτυξη των μικρών νεοπαγών εταιρείων. Δεύτερον, χαιρετίζω αυτό που είπατε για την απλούστευση όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδοτική στήριξη, αλλά ε, πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποίηση ανάμεσα στις επιδοτήσεις και, και τα δάνεια που δίνονται. Πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω αυτό το θέμα. Επίσης, συμφωνώ με τον κύριο Χέιλερ για, για τα σχόλιά του για την κοίηση. Τώρα, για την Βρετανική θέση. Πρώτον, ακαδημαϊκοί ερευνητές. Εκεί πραγματικά έχουμε πάρα πολλά στοιχεία για το ότι αποκλείονται και πρέπει να εξασφαλιστεί ότι θα ε, ε, ε, διατηρηθεί η χρηματοδότηση όσο είμαστε ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερο για το JET και το ITER και για την αναγκαιότητα που υπάρχει για το JET όσον αφορά το μέλλον του ITER. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Λεοπρόεδρος. Να σας συγχαρώ και εγώ για την νίκη του Μάρη στο Wimbledon. Συνάδελφος Μπλάνκο Λόπες. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκαν κάποιες ε, ε, μελέτες που είχαν ε, ορίσει κάποιες επιτροπές μεταξύ των οποίων και η δικιά μας σχετικά με την αποτίμηση και το, της προετοιμασίας για τον ορίζοντα 2020 υπάρχουν στοιχεία καλά και στοιχεία αρνητικά. Αρνητικά βεβαίως έχουν ταυτιστεί, έχουν ταυτοποιηθεί συγγνώμη, σε σχέση με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες λοιπόν επιχειρήσεις δεν έχουν σωστά, ε, ε, σωστές πληροφορίες σχετικά με τα ισχυρά ε, ή όχι σημεία τους και το ποσοστό επιτυχίας είναι γύρω στο 6%. Είναι πάρα πολύ χαμηλό και επίσης η δυνατότητα άντλησης χρηματοδότησης προγραμμάτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν είναι υψηλό. Έχετε ταυτοποιήσει τα πρόοδο προβλήματα αυτά κύριε Επίτροπε και κάνετε κάτι έτσι ώστε να τα ξεπεράσετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Πρόεδρε, λέει η κυρία Μερσέντες. για το άρθρο 161, στα πλαίσια του άρθρου 161 για την ε, συνεργασία είχαμε υποβάλει μια μεγάλη πρόταση ε, επιστημονικής αλλά και διπλωματικής ε, συνεργασίας όσον αφορά την τροφοδότηση σε νερό συγκεκριμένων περιοχών. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και πρέπει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Επίσης, ε, από ό,τι μαθαίνουμε, ενδεχομένως ε, ε, θα προσθεθούν εδώ και στο ίδιο πρόγραμμα και κάποια στοιχεία για τη μελέτη των μεταναστευτικών ροών, αλλά αυτό ίσως δυναμητήσει το όλο πρόβλημα και δυσκολέψει και την έγκρισή του. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να το μελετήσετε αυτό, γιατί δεν είναι δυνατόν να δυναμητιστεί ή να τεθεί σε κίνδυνο μια, κατά την άποψή μου, θεμελιώδου σημασία προτεραιότητα. Όσον αφορά τον ορίζοντα 2020 και την ενδιάμεση αξιολόγηση, εγώ θα ήθελα ε, να διευκρινιστούν κάποια στοιχεία ε, να μας πείτε δηλαδή εδώ στην Επιτροπή Ήτρε πώς, προχω... πώς προτίθεστε να προχωρήσετε, ποια είναι τα στοιχεία τα οποία έχετε κατανοήσει ότι δεν είναι σωστά και που θα πρέπει να τα τροποποιήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πίτροπε. Χαίρομαι που σας βλέπω και πάλι εδώ. Όταν μιλούμε για καινοτομία, νομίζω ότι είναι πάντα σημαντικό να υπογραμμίζουμε τον ρόλο της βασικής ε, έρευνας, γιατί ξέρουμε αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε καινοτομία. Και βεβαίως επενδύσει για τις υποδομές, ερευνητικές υποδομές, πολύ σημαντικό τμήμα της ε, βασικής έρευνας. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία λοιπόν που μας παρουσιάσατε είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Θα ενταχθεί στην ενιαία ψηφιακή αγορά και στην ε, αγορά μας ε, που κατευθύνεται με βάση τα δεδομένα. Έχω ορισμένες ερωτήσεις, θα πείτε και εσείς ποια είναι η γνώμη σας. Τώρα που θα θεσπίσουμε αυτό το νέο ανοιχτό ε, νέφος, είναι πολύ σημαντικό θεωρώ να βασιστεί σε υφιστάμενες υποδομές και στις αρμοδιότητες που έχουμε να εντοπίσουμε κενά και να τα καλύψουμε και σε υπηρεσίες ε, που εξυπηρετούν τον χρήστη. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε τι υφιστάμενε υποδομέ κατά το δυνατόν και τι ικανότητε και αρμοδιότητε που ήδη διαθέτουμε. Μετά για το μοντέλο χρηματοδότηση. Βλέπω ότι ακόμα μένει ανοιχτό το πώ ακριβώ ε, θα γίνεται η χρηματοδότηση του ερευνητικού νέφου, επιστημονικού νέφου, όμω θα πρέπει να βρούμε ένα βιώσιμο χρηματοδοτικό μοντέλο και οι ε, ρόλοι και οι ευθύνε θα πρέπει να διευκρινιστούν. Από πλευρά κρατών μελών, από ό,τι βλέπω, θα υπάρχει συμμετοχή ε, και χρηματοδότηση. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχουν και εθνικά ωφέλη, κατά τη γνώμη μου. Θα ήθελα να πείτε δύο λόγια παραπάνω για το πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ε, υφιστάμενε υποδομέ και τι είδου χρηματοδοτικό μοντέλο θα έχουμε. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Έλερ, θέλετε να επανέλθετε πολύ, πολύ γρήγορα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Για το Brexit, Υπάρχει αυτή η παρανόηση από κάποιου ότι ε, παίρνουν περισσότερα από ό,τι δίνουν ή το αντίστροφο. Τέλος πάντων, για το, την επίκριση του άρθρου 50 λέτε ότι θα έχουν δύο χρόνια, αλλά αυτό ήδη συνδέεται με το νέο 2020. το πρωτόκολλο Ευρατόμ θα πρέπει να παραταθεί του χρόνου. Και αυτό συνδέεται άμεσα με τον Βασίλειο. Από τεχνική σκοπιάς λοιπόν, είναι ρεαλιστικό να πούμε ότι υπάρχει αυτό το χρονοδιάγραμμα των δύο ετών, γιατί υπάρχουν πολλά ακόμα ζητήματα που επήγουν και δεν μας δίνουν το χρονικό περιθώριο που προβλέπεται από το άρθρο 50. Ο Πρόεδρος, να προσθέσω κύριε Επίτροπε, στο τέλος αυτού του γύρου ερωτήσεων, στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Συμβουλίου δεν θεσπίστηκε κανένας καινούριο θεσμό. Χρηματοδοτούμε την θεμελιώδη βασική έρευνα. Δεν είχαμε τέτοιου είδου έρευνα σε τέτοιο βαθμό στο 7ο πρόγραμμα, συγγνωμη πρόγραμμα πλαίσιο. Ξεκίνησε το 7ο. Και ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη, γιατί όλη αυτή η έρευνα διεξήχθη στα Ινστιτούτα δεν ήταν μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων στο ERC. Αλλά οδήγησε σε τεράστια ε, προαγωγή της ευρωπαϊκής έρευνας σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Καινοτομίας. Το... Για το Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας. Σε αυτή την περίπτωση, ούτε εδώ διαμορφώσαμε ένα νέο θεσμό υπήρξε μια δικτύωση μεταξύ υφιστάμενων θεσμών. Ήταν πολύ ωφέλιμο λοιπόν ε, να συμβάλλουν όλοι αυτοί ε, στην έρευνα από κοινού και με την ε, βιομηχανία μας. Έχω το ίδιο ερώτημα λοιπόν και εδώ. Δεν θα υπάρξουν νέες δομές από ό,τι βλέπω. Ούτε ας πούμε θα τους δοθεί κτίριο, για παράδειγμα στο EIC. Τι συμβαίνει με τον προπολογισμό. με πολύ απλά λόγια το ρωτώ. Μπορεί να υπάρχει προπολογισμό, αλλά θα πρέπει να ε, βοηθήσει αυτό ο προπολογισμό, αυτή η χρηματοδότηση, να βοηθήσει οι φυστάμενε δομέ να είναι πιο αποδοτικέ, όπω κάναμε και στι προηγούμενε περιπτώσει που προανέφερα. Δεν αντιβαίνουμε λοιπόν ούτε στους, ε, στα ευρωπαϊκά όργανα, ούτε στην ευρωπαϊκή βιομηχανία. Του βοηθήσαμε. Έχουμε λοιπόν ενδεχομένω χρηματοδότηση, ίσω και όχι. Αν όμως δοθεί χρηματοδότηση, πώς θα δοθεί, ούτω ώστε να μην αντιβαίνει, να μην ανταγωνίζεται όλες τις υπόλοιπες δομές που ασχολούνται ακριβώς με την καινοτομία. Very Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω από εσάς. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. η προαγωγή της ευρωπαϊκής έρευνας και το branding που προέκυψε από το ERC, που θεωρώ ότι είναι πραγματικά σημαντικό. Πρέπει και για την καινοτομία να δώσουμε αυτή την εικόνα, την προβολή αυτής της εικόνας, του branding, όπως κάναμε στην τομέα της έρευνας. Συμφωνώ. Από την αρχή όμως η πρόθεση ήταν να βρούμε κάτι που να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή ακόμα και χωρίς χρηματοδότηση. Δηλαδή, αν αυτές οι προτάσεις λειτουργήσουν και χωρίς χρηματοδότηση, είναι εξαιρετικές ιδέες. Αν χρειαζόμαστε χρηματοδότηση για να τις υλοποιήσουμε, δεν είναι και τόσο τρομερές. Προς το παρόν, λοιπόν, Το μοναδικό που χρειάζεται χρηματοδότηση από αυτά τα δέκα, που προανέφερα είναι η δημιουργία τη συμβουλευτική ομάδα. Όμω, προ το παρόν, έχουμε ιδέε ε, που έχουν ε, σχέση με τη μεθοδολογία μας και πώς ε, καταπιανόμαστε με τις πρωτοβουλίες μας. Θα το δούμε λοιπόν αυτό. Προς το παρόν λοιπόν οι αλλαγές αυτές δεν συνδέονται με τον προπολογισμό αυτή τη χρονική στιγμή. Αν δείτε όμως και τον προπολογισμό με όλα τα μέσα που έχουν στη διαθεσή μας αυτή τη στιγμή, βλέπετε ότι ήδη υπάρχει ένας ε, σημαντικός προπολογισμός γι' αυτό. Αυτό εναπόκειται και στο Κοινοβούλιο για να μας δώσετε και περισσότερες ιδέες. Όμως αυτό θεωρήσαμε ότι θα ήταν μια καλή ιδέα ακόμα και χωρίς προπολογισμό, αλλά θα δούμε. Μετά περνώ στις άλλες ερωτήσεις. Πόσο έχω, 10 λεπτά. Ο κύριος Ζανονάτο. Το ερώτημα για την πρίμα το έθεσε και ο κύριος Ζανονάτο, η κυρία Καστίλιο Βέρα και η κυρία Καπεθόν Ρουίθ. Λοιπόν, για την πρίμα, λοιπόν, ξέρετε ότι εγώ είμαι αναφαντών υπέρ αυτού του προγράμματος και προσωπικά έχω ασχοληθεί με, όλα, με το πρίμα. Οριστικοποιούμε αυτή τη στιγμή την αξιολόγηση αντικτύπου. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα στη Γενική Διεύθυνση που ασχολείται με αυτό το θέμα. Υπήρξε ε, και άτομο από, σε επίπεδο μάλιστα γενικού διευθυντή Τρομερή λοιπόν συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα. Ε, η διυπηρεσιακή διαβούλευση θα λάβει χώρα το καλοκαίρι και μετά θα περάσουμε στην ε, υιοθέτηση τον Οκτώβριο. Θα περάσει στο Κοινοβούλιο και Συμβούλιο για την νομοθετική διαδικασία. Προς το παρόν ε, δεν μπορώ να σας πω και πολλά, γιατί η διαδικασία είναι εν εξελίξη και δεν μπορώ, δεσμεύομαι δηλαδή και από κανόνες εμπιστευτικότητας. Ξέρουμε όμως ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα για το μέλλον. Ας ξεχάσουμε το όνομα πρίμα. Πρόκειται για την τροφή και το νερό στη Μεσόγειο. Κάποιες φορές το ξεχνάμε. Κύριε Καστιγιοβέρα. το σχόλιο σας σχετικά με την ανάγκη επιτάχυνσης ε, του προγράμματος ε, για το νέφος. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Είναι απαραίτητο και για τους ερευνητές ε, και για τους ε, ε, και για τους επιστήμονες ε, και στην Ευρώπη. Και αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που μου κάνουν οι ερευνητές και οι επιστήμονες. Πότε θα έχουμε αυτό το νέφος. Αυτό και άλλωστε και προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να προχωρήσει πολύ, αλλά υπάρχουν και διαδικασίες τις οποίες πρέπει να διατηρήσουμε. Μετά. Ο κύριος Ζωρίνιο πήρε το λόγο στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως γνωρίζετε, όταν μιλούμε για αποδέσμευση τοξικών ουσιών, ε, δεν μπορώ να πάρω θέση για το ERC. Πάντως είναι μια κατάσταση που παρακολουθούμε και το συνεγγύς υπάρχει αυτή η ομάδα επιστημόνων και εμπειρογνωμόνων που μελετά ακριβώ το θέμα των εκπομπών. Μία από τις πρώτες δραστηριότητες που ανέλαβαν ήταν αυτή. Θέλουμε πραγματικά να το μελετήσουμε σε βάθος. Πρόκειται για πραγματικό επιστημονικό συμβούλιο που ε, μας βοηθάει. Τα έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Είχα τη δυνατότητα να μιλήσω και με τον αρμόδιο υπουργό της Πορτογαλίας. Ξέρω ότι υπήρξε θέμα με τις Αζόρες και με τη στρατιωτική βάση και κατά πόσο οι Αμερικανικές αρχές ε, θα ε, αποχωρούσαν. Επί της ουσίας, ε, με αυτό το πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει στην το 2020, αλλά θα δούμε. Ευχαριστώ. Μετά, ένα ερώτημα και σχόλιο μαζί από τον κύριο Μπόνι για την ε, εμπλοκή, τη συμμετοχή των Ευρωπαίων επιστημόνων στο επιστημονικό νέφος. Ναι, η προσέγγιση πρέπει να είναι από τα κάτω προς τα πάνω. Να δούμε τι ακριβώς χρειάζονται και θέλουν οι επιστήμονες για το μέλλον. Οπότε σε κάθε περίπτωση εμείς θα διαβουλευτούμε με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να γνωρίζουμε ποιες ε, είναι οι υπηρεσίες που χρειάζονται στο data mining. Είναι πράγματι πολύ εύστοχο το σχόλιο που κάνατε λοιπόν. Μετά, η κυρία Βίνικ. Ε, σας καλωσορίζω κι εγώ και σας εύχομαι κάθε επιτυχία εδώ στο έργο σας. Για το risk capital με ρωτήσατε. Εμείς ε, είμαστε υπέρ του να δημιουργηθεί ένα ταμείο των ταμείων στην Ευρώπη. Ε, θέλουμε να δημιουργηθεί ένα ταμείο ιδιωτικής διαχείρισης με δημόσια κονδύλια και ιδιωτικά κεφάλαια μεταξύ μισού και ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Αλλά μαζί με ιδιωτικά κεφάλαια, γιατί αυτά χρειαζόμαστε προκειμένου να γίνει αυτή η κλιμάκωση, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Αυτό κάνουμε λοιπόν σε αυτόν τον τομέα, μιας και με ρωτήσατε, και ελπίζω να έχουμε και άλλες ευκαιρίες για το πώς μπορούμε να έχουμε και άλλες ευκαιρίες συζήτηση για το πώς μπορούμε να άρουμε τους περιορισμούς και τα εμπόδια και να πλουστεύσουμε τις διαδικασίες. Δική μας πρόθεση πάντως είναι σε κάθε περίπτωση να αξιοποιήσουμε και την Ολλανδική εμπειρία σε αυτόν τον τομέα. Πράγματι ήταν πολύ σημαντικά αυτά που αναφέρατε. Μετά. Κύριε Λιμπάξα, για τον διαχωρισμό. Γνωρίζετε τη σημασία που αποδίδω σε όσα σχετίζονται με την διεύρυνση, την δικτύωση και την προεδρία της ε, Ευρωπαϊκής, ε, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας. Εμείς θέλουμε να κάνουμε όσο, ό,τι γίνεται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και θέλουμε να τα εμπλέξουμε στην στελέχωση και την δικτύωση. Ε, θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε αυτήν τη διάσταση. Θα συνεργαστώ και με τη συνάδελφή μου την ε, κυρία Κορίνα Κρέτσου για αυτόν τον τομέα. Κοιτάξτε, θα ήθελα να σας πω ότι και σε αυτή την περίπτωση, ε, για την περίπτωση της Ελβετίας, το μπαλάκι είναι από την πλευρά της Ελβετίας. Εγώ Βεβαίως προσυπογράφω ότι, ότι η έρευνα στην Ζηρίχη, στην Ελβετία είναι παγκοσμίω, γνωστή και αποδεκτή, αλλά βεβαίως τα περαιτέρω θα εξαρτηθούν ε, και από τις συμφωνίες που έχουμε κάνει ε, με την ε, ε, Ελβετία ευελπιστώ ότι θα ε, συνεχιστεί η ε, έρευνα και η συνεργασία με την πολύ σημαντική ελβετική έρευνα. Μετά ένα ερώτημα από την κυρία Μούντι για όλα όσα σχετίζονται με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ελπίζω εγώ θα βρεθώ σύντομα στο Μάνσεστερ και θα το πω και στους ανθρώπους εκεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι τα πράγματα μένουν ως έχουν προς το παρόν. Έχετε τις υποχρεώσεις σας, τα δικαιώματά σας και αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι η ερευνητική κοινότητα, η επιστημονική κοινότητα πρέπει να συνεχίσει στο δρόμο που έχει χαράξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θέλω λοιπόν να ε, τροφοδοτήσω αυτή την παραφιλολογία ότι κάποιοι θα αποκλειστούν και κάποιοι θα ωφεληθούν Σκοπός μου είναι ολόκληρη η επιστημονική κοινότητα να ε, ωφεληθεί. Έχω μιλήσει και με τον κύριο Τζόνσον, τον Υπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου και μου έχει, με έχει ενημερώσει ε, για το ότι φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια τέτοια φαινόμενα. Χρειάζομαι όμως στοιχεία. Ε, θα συνεχιστεί η συζήτηση αυτή, σας διαβεβαιώ. Μετά, άλλα τρία θέματα που θέλω να απαντές, οποία θέλω να απαντήσω. Για τις μικρομεσαίες ρώτησε ο κύριος ε, Μπλάνκο Λόπες. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καινοτομίας μπορεί να απαντήσει στην ερώτησή σας. Ας πούμε, αυτό που με ρωτήσατε για την αξιολόγηση. Πιστεύω ότι θα πρέπει όταν κάνουμε αξιολόγηση ενός μιας μικρομεσαίας, θα πρέπει να είμαστε ε, πρόσωπο με πρόσωπο το κατά πόσον ε, θα μπορέσουμε να κάνουμε αλλαγέ και ο τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι αλλαγέ αυτέ, ε, ε, βεβαίω μα απασχολεί αυτό. Επίση, συνεχίζω στα Ισπανικά για την κυρία Καπεσόν Ρούγε. Για το πρώτο σα απήντησα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα όντως εμείς πρέπει να δούμε μέχρι το 2017 ε, πώς θα κάνουμε τη διαβούλευση με τους εμπλεκομένους ε, και βεβαίως θα ε, λάβουμε και όλες τις πληροφορίες ε, τις οποίες μας έχετε δώσει και σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω γι' αυτό. Έχουμε μιλήσει ήδη μεταξύ μας για το θέμα αυτό και ευελπιστώ ότι στο τέλος του 2017 θα έχουμε την δυνατότητα, έχοντας ε, ε, όλη αυτή την πληροφόρηση, να μπορέσουμε να κάνουμε και την ανακοίνωση για το νέο πρόγραμμα και την νέα αξιολόγηση. Και μετά, συμφωνώ με τα σχόλια της κυρίας Βιλκούνων ήταν πολύ θετικά σχετικά με την υποδομή και την διαλειτουργικότητα και για αυτό που είπε ο κύριος Χέλε, για τα ερωτήματα που έθεσε, τα οποία είναι πολύ σημαντικό, σημαντικά. Όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι μεγάλο το ερώτημα αυτό που θέσατε για την Ευρατόμ. Ε, εγώ θα δουλέψω νυχθημερών για να λύσουμε αυτά τα θέματα 24 ώρες το 24ωρο ε, σας διαβεβαιώ, αλλά βεβαίως είναι σίγουρο ότι αυτό το ζήτημα είναι τεράστιο και θα μας απασχολήσει το επόμενο διάστημα. Αυτά είχα να πω κύριε Πρόεδρε, από την πλευρά μου. Um, Κάτι διαδικαστικό. Έθεσα πέντε ερωτήματα σχετικά με την ανοιχτή πρόσβαση και την ανοιχτή επιστήμη προς την Κομισιόν γιατί μου υπόθηκε ότι υπάρχει αυτός ο νέος κανόνας ότι μπορούν οι ευρωβουλευτές να θέσουν έως και πέντε γραπτές ερωτήσεις. Δεν το ήξερα γιατί παλιότερα είχα θέσει και περισσότερα ερωτήματα. Θα ήθελα λοιπόν να ε, με διαβεβαιώσει ε, ο Πρόεδρος ότι αυτό όντως ισχύει. Γιατί αν ισχύει ε, πρόκειται για σοβαρό περιορισμό των δυνατοτήτων του κοινοβουλευτικού ελέγχου ε, νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ κάποια επίσημη πολιτική ή τέτοια απόφαση. Ε, νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποφασίσει σε διοικητικό επίπεδο γιατί ε, στην ουσία περιορίζεται και το δικαίωμά μας στο να θέτουμε ερωτήσεις. Επίσης να σε ευχηθώ καλό καλοκαίρι και να ευχαριστήσω και εγώ τους δερμηνείς. Πρόεδρος, θα το ε, διερευνήσω το θέμα που εγείρατε. Είναι πραγματικά σημαντικό να γνωρίζουμε με ακρίβεια τι συμβαίνει. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Θα τα πούμε στην επόμενη ε, συνεδρίαση, συνάντησή μας. Σας εύχομαι να έχετε εκπληκτικές διακοπές, να παίξετε και λίγο ε, ποδόσφαιρο αν μπορέσετε με τα παιδιά σας. Τι έχετε, αγόρι κορίτσι. Ένα και ένα. Βεβαίως. Λοιπόν, και οι γυναίκες παίζουν εξαιρετικό πελέσφαιρο. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την παρουσία σας εδώ. Συνάδελφοι. Θα ξαναλέμε στις 3 για την τελευταία συνεδρίασή μας. 3 το απόγευμα. Είστε όλοι ε, προσκεκλημένοι. Θα μιλήσουμε με την Σλοβακική Προεδρία από την αρχή. Θα λέμε σε 2,5 ώρες.